Good afternoon, gentlemen. evening already. Can we... Λοιπόν, αν την καλοσύνη, ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Είναι πολύ σύντομη η ημερήσια διάταξη. Είναι έκτακτη συνεδρίαση. Έχετε κάποιες προτάσεις, μήπως έχετε κάποια σχόλια για την ημέρησια διάταξη. Όχι, εγκρίνεται λοιπόν. Δεν έχω κάποιες ειδικέ ανακοινώσεις για την ε, Περιφερειακή Επιτροπή. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το βασικό θέμα μας για σήμερα, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βάλτις Ντομπρόφσκης, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για το ευρώ και το κοινωνικό διάλογο σχετικά πρόταση επιτροπή για την κατάρτιση ενό προγράμματο στήριξη των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020. Το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πρόταση για έναν κανονισμό για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα στήριξη των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 με 2020. Πρόθεση του προγράμματος αυτού, διαθωτικών μεταρρυθμίσεων, στήριξης αυτών, είναι να εφαρμόσουν θεσμικές, διοικητικές και διαθωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και βοήθεια για αποτελεσματική χρήση των πόρων της ενώσεως για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η θέση απασχόλησης. Θα, παρασχεθεί συγγνώμη υποστήριξη κατόπιν ετοίμας των κρατών μελών και κατόπιν συστάσεων κατά χώρα που θα εκδίδονται σε σχέση με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τα προγράμματα οικονομικής ε, αναδιάρθρωσης ή βάση των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη κατόπιν ιδέας πρωτοβουλίας. Η πρόταση έχει το άρθρο 175 σαν νομική βάση και το άρθρο 197 μια δυτή ε, νομική βάση και συναπάγεται τροπολογία του κανονισμού με τις κοινέ διατάξεις. Προτείνεται ότι το ο προπολογισμό των 142,8 εκατομμυρίων για την πολιτική περίοδο, προπολογισμό, θα αφαιρεθεί από τον προπολογισμό τεχνική αραγή που είναι στη διάθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το ERDF, ESF και το Ταμείο Συνοχής. Κοινωνικό Ταμείο και περιφερειακή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος να συζητηθούν οι αρμοδιότητες για αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά στις Μαΐου του 2016 η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε περί της κατανομής των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων επιτροπών για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας θεωρήθηκε ότι είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θα ετοιμάσει μια συν, ε, ε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Στερικού Κανονισμού, η Επιτροπή Προπολογισμού θα, ε, θα κινηθεί σύμφωνα μετά το 53 συν οι επιτροπή Κολτ και Πέτς θα, θα παράξουν τις γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 53. Μετά από τις αποφάσεις αυτές ξεκινάει η εργασία μας και συγκάλεσα τη σημερινή έκτακτη σύνοδο μας ούτως ώστε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Βάλτης Ντομπρόσκης, να παρουσιάσει μια πρόταση στην, ε, στην Επιτροπή μας και τους οι των γνωμοδοτήσεων των διαφόρων επιτροπών που προανέφερα. Έχουμε τους συνεισηγητές μαζί μας. Αποφασίσαμε να έχουμε συνεισηγητές για αυτό το θέμα. Την κυρία Κρέλ και τον κύριο Βαν Νίστελ Ρόι. Και έχουμε και σκιώδεις εισηγητές παρόντες στην αίθουσα και εισηγητές από άλλες επιτροπές, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Εισηγητής είναι ο κύριος Σογκόρ. Σωστά, σας Σωστά προφέρω το όνομα σας. Αρκετά. Εντάξει. Πλησίασα. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Προπολογισμών, η συγγητής, ο κύριος Γιάνν Όλμπρεχτ, είναι παρόν. Καλώς ήρθατε. Δυστυχώς, ο εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων δεν έχει ακόμα διοριστεί. Αλλά μέχρι το τέλος του μηνός θα γνωρίζουν ποιος θα είναι, ίσως την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Ελπίζω αυτό το μήνα, ελπίζω. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Ντομπρόσκης, να προβεί στην παρουσίασή του και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη μας για σχόλια, για ερωτήσεις, ξεκινώντας από τους συνεισηγητές, τους εισηγητές των άλλων επιτροπών και τους κοιόδης εισηγητές. Κύριε Ντομπρόσκης, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να έρθω να συζητήσουμε την υποστήριξη των διαθωτικών μεταρρυθμίσεων και το σχετικό πρόγραμμα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις συστάσεις κατά χώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συστάσεις για την εφαρμογή διαθωτικών μεταρρυθμίσεων, για τον εξυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών, να ενθανηθούν οι επενδύσεις, να αυξηθεί, αυξηθούν θέσεις εργασίας και να προωθηθεί η σύγκληση εντός των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι οι μεταρρυθμίσεις λειτουργούν τα κράτη-μέλη εκείνα που ήδη εφάρμοσαν φιλόδοξα μεταρρυθμιστικά προγράμματα όπως η Ισπανία, Ιρλανδία, η Πορτογαλία, τα βαλτικά κράτη πριν από αυτό, τώρα αυτά τα κράτη ε, καλύπτουν τη διαφορά και πολλά από τα κράτη έχουν πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, τους υψηλότερους και αυτό μεταφράζεται σε θέση απασχόλησης, λιγότερη φτώχεια και λιγότερο κοινωνικό αποκλεισμό. Όμως, κατά μέσο όρο, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων δεν είναι ικανοποιητική. Η παρούσα αξιολόγησή μας είναι εξής, ότι τα κράτη-μέλη είναι μεταξύ περιορισμένης και κάποιας προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των καταχώρα συστάσεων και των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Σαφώς παραδεχόμαστε ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι κάτι που απαιτεί πολιτικό θάρρος για να αντιμετωπιστούν καμιά φορά ισχυρά συμφέροντα. Και κάποιες μεταρρυθμίσεις κοστίζουν δημοσιονομικά και κάποιες μεταρρυθμίσεις ίσως είναι περίπλοκες από τεχνική σκοπιά και πολύ συχνά οι χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά διοικητικό και θεσμικό δυναμικό η νομοθεσία δεν αρκεί. Αυτό που μετρά είναι η σωστή εφαρμογή και υλοποίηση και πολύ συχνά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Για να υποστηριχθούν τέτοιες χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε, κινείται ενεργά και πέρσι δημιουργήσαμε μια υπηρεσία για υποστήριξη εθωτικών μεταρρυθμίσεων και υποβάλαμε μια πρόταση για συγκεκριμένο πρόγραμμα, εργαλείο μάλλον, για υποστήριξη των, μεταρρυθμιστικών, των μεταρρυθμίσεων αυτών, των διεθωτικών και σχετικό πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος αυτού, της στήριξης των μεταρρυθμίσεων, είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, κυρίως στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, κυρίως σύμφωνα με τις συστάσεις κατά χώρα και τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, όπου εκεί η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κάτι παίζει ρόλο, ή η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που βοηθούν την ανάπτυξη. Από τη στιγμή που αυτά τα άλλα μέτρα αρθιγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το πρόγραμμα θα προβλέπει και βοήθεια για αποτελεσματική χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πιο συγκεκριμένα βέβαια τα ευρωπαϊκά διαθωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδυτικά και θα μπορούν να συμμετέχουν και τα 28 κράτη-μέλη εφόσον το ζητήσουν. Το φάσμα των διαφόρων τομέων πολιτικών που είναι επιλέξιμη για υποστήριξη ε, θα είναι ευρύ φάσμα από αποτελεσματικές δημόσιες λειτουργίες, οικονομική διαχείριση, διαχείριση των εσόδων, Αγορά εργασία, κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές για ανάπτυξη, για επιχειρηματικότητα και πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η υποστήριξη θα παρέχεται άμεσα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και από εξωτερικούς παρόχους, εκείνους που ασχολούνται με το θέμα σε αλλα κράτη-μέλη ή ειδικευμένου διεθνείς οργανισμούς. Θα τονιστεί ιδιαίτερα η πρακτική υποστήριξη, η επιτόπια, κατάρτιση ε, επιτόπου την ώρα της δουλειάς αντί να γίνονται μαθήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τα υποστηρικτικά μέτρα σε στενή συνεργασία με τα κάτι μελη που ενδιαφέρονται βάσει με το αρχικό τους αίτημα και κατόπιν αναλύσεως της επιτυχίας. Η υποστήριξη θα είναι αμοιβαία συμφωνία μεταξύ κράτους μέλους και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε θα ενστερνίζεται το πρόγραμμα το κράτος μέλος και συμμετέχει πιο πολύ. Εξυπακούεται βέβαια ότι η επικάλυψη των προσπαθειών και της χρηματοδοτήσεως είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί. Θα εξασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη σύμφωνα με, τα, με αυτό το σύστημα θα συμπληρώνει άλλες δράσεις, δημιουργία δυναμικού και τεχνική βοήθεια που σχετίζονται με άλλα προγράμματα και σύμφωνα με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και τεχνική βοήθεια και άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από ε, ταμεία όπως είναι το κοινωνικό ταμείο. Συμπληρωματική λειτουργία λοιπόν. Λοιπόν, αυτό, πώς θα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό στήριξης διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Θα έχουμε συγκεκριμένο κονδύλι για ένα πρόγραμμα που θα είναι στα 142,8 εκατομμύρια ευρώ ε, για την επόμενη τετραετία, δηλαδή 2017 μέχρι το 2020. Αυτό το ποσό θα προέρχεται από αναδίπλωση ε, των πόρων για τεχνική αρρωγή που κεντρικά είναι στη διάθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα ταμεία για την πολιτική συνοχή και τους πόρους για την άπτυξη της υπαίθρου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης τεχνικής αρρωγής και των πόρων που είναι διαθέσιμοι για όλα τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με την συγκεκριμένη διανομή πόρων τα Ταμεία Συνοχής και του Ταμείου Αναπτύξης Υπέθρου όλα αυτά θα παραμείνουν αμετάβλητα. Δηλαδή δεν πειράζουμε καθόλου τα εθνικά πλαίσια. Σχετικά με αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισαν ποιο είναι το ποσό που θα χρηματοδοτείται αυτό το πρόγραμμα, λαμβάνοντα υπόψη τι αναμενόμενε ανάγκε για την ε, υλοποίηση τη τεχνική αρρωγή και των δράσεων σύμφωνα με την πολιτική συνοχή και την πολιτική για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Επιτρέψτε μου να επιθυμίσω ότι την περίοδο 2014-2020 έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα διαθέσιμα για τεχνική αρρωγή κάτω από τα πλαίσια των τεσσάρων ταμείων, του ERDF, ESF, του Ταμείου Συνοχή και του Ταμείου για την Ανάπτυξη Πέθρου, Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Περιφερειακή ανάπτυξη. λοιπόν. Λοιπόν, αυτά είναι συγκρίση με, τα προηγούμενα, με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 400 εκατομμύρια είναι η αύξηση όσον αφορά την κεντρική τεχνική αρρωγή που παρέχεται σε αυτή την περίοδο. Και η ανάλυση μα τι καταδεικνύει, ότι ακόμα και μετά από την αναδιάταξη την αντίπλωση των πόρων θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τεχνική αρρωγή κατόπιν πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συγκρίση με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013. Κάθε χρόνο οι αρχέ του προπολογισμού εξετάζουν το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί συμπεριλαμβάνεται και μια αιτήσια κατανομή για αυτό το πρόγραμμα που συζητάμε. Τέλος, τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση, αν το επιθυμούν, να μεταφέρουν τους πόρους τους από τα εθνικά τους κονδύλια για την τεχνική βοήθεια στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου, σε αυτό το πρόγραμμα συζητούμε, για να, έχουν τεχνική αρρωγή. Για το διευκολύνουμε αυτό, κάποιες τροποποίησεις των κοινών του, του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις και του, του κανονισμού για το, το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης χρειάζονται να τροποποιηθούν Λοιπόν, ελπίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για την υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η οικονομική τους ανάκαμψη, να, να ισχυροποιηθεί δυνατότητα προσαρμογής και να προωθήσουμε την σύγκληση εντός κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε το πρόγραμμα αυτό και να προωθήσετε γρήγορα την νομοθετική διαδικασία, τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν από την υποστήριξη από τον Ιανουάριο του 2017, όπως ε, αρχικά είχε προγραμματιστεί στην πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη βέβαια να σας βοηθήσει ε, σε αυτή τη δουλειά και να σας δώσει και τις αναγκαίες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στις απόψεις σας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Φανίστελρο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, όσοι εισηγητές για... δουλεύουμε ως ομάδα για την κοινή νομοπαρασκευαστική διαδικασία και θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλήσατε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να περιβάλλει αυτή την πρόταση. Αλλά και για τα απαραίτητα κονδύλια. Το σημαντικό είναι να κινηθούμε γρήγορα και να σχεδιάσουμε να προγραμματίσουμε σωστά τη δουλειά μας. Η πρόεδρος της Επιτροπής έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα εργασιών μας και αυτό σημαίνει ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να συνδυαστεί, να συντονιστεί, να προχωράει το έργο σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Είναι καλή αυτή η πρώτη συνάντηση για να έχουμε τις πρώτες πληροφορίες και χαιρόμαστε ιδιαίτερως διότι η Επιτροπή Προεπολογισμού έχει ήδη εισηγητή ε, ο οποίος είναι παρόν και ο εισηγητής της ε, Επιτροπής Απασχόλησης είναι παρόν για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ενώ και οι λοιπές επιτροπές ΠΕΣΟΥ και ΚΟΥΛΤ έχουν ορίσει εισηγητές για την έκδοση γνωμοδότησης. Η Επιτροπή Οίκων εντάσσεται στον κανόνα 54. Δεν υπάρχει ακόμα εισηγητής από πλευράς ΕΙΚΟΝ. Ξέρω ότι επιθυμούν να στηρίξουν την πρότασή σας και γι' αυτό γρήγορα θα ανακοινώσουν τη θέση τους και θα μπορέσουμε όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να ε, ε, επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας. Σε σχέση με το προγραμματισμό που συζητήσαμε χθες, να σας πω ότι βεβαίως και θα μπορούμε να έχουμε ένα προσχέδιο έκθεσης πριν από το καλοκαίρι, θα μπορέσει να σταλεί για μετάφραση μέχρι τις 15 Ιουλίου πριν την διακοπή του Αυγούστου θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το προσχέδιο έκθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου συνεργαζόμενοι καταλήλως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι η εβδομάδα μετά τις 14 Σεπτεμβρίου και στις 11 Οκτωβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες σε συνεδρίαση, ενώ θα ψηφίσουμε την έκθεση τον Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή και αγαστή συνεργασία, κυρίως με την Επιτροπή ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα θα πρέπει να πάει η έκθεση πριν τα τέλη της χρονιάς στην Ολομέλεια. Έτσι κάπως ε, σκεφτόμαστε να δουλέψουμε. Και αν οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ ε, επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα ε, και οι ίδιε για τη δική του έκθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε και να το πετύχουμε. Είμαστε συνομοθέτε και θα πρέπει ο κανονισμός να προσαρμοστεί. Και έτσι μπορούμε να ενσωματώσουμε όλες τις απόψεις. Δηλαδή μπορεί να λυθεί το θέμα μέσα στο 2016. Θα ήθελα να κάνω ένα, το εξή σχόλιο. Υπάρχουν τα χρήματα από την τεχνική βοήθεια και τις επενδύσεις και τα παίρνετε από εκεί είναι διαθέσιμα τα κονδύλια. Είπατε ότι δεν επηρεάζονται αυτοί οι χρηματοδοτικοί φάκελοι. Γίνεται άλλη ιεράρχηση. Μεταφέρονται στην Ένωση τα κονδύλια με την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας λέτε δύο λόγια παρακαλώ για το τι αντίκτυπο αυτό θα έχει στην περιφερειακή πολιτική. Είναι χρήματα δωρεάν, δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπο στην περιφερειακή πολιτική. Ελεύθερα μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περί τίνος πρόκειται. Και δεύτερο ερώτημα. Αυτά τα χρήματα στα οποία αναφερθήκατε ε, είναι το σύνολο, είναι όλα τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για όλη την προγραμματική περίοδο ή του χρόνου θα επανέλθετε με επόμενη πρόταση και ε, δύο χρόνια μετά με επόμενη και ούτω καθεξής. Έχει γίνει αναδιοργάνωση επίσης στο επιτελείο σας, στις υπηρεσίες σας. Πώς αυτό θα λειτουργήσει. Υπάρχουν δεσμεύσεις των κρατών μελών πιστώσεις, μάλλον οι χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο δεν θα υποβάλουν αιτήματα. Οπότε πώς θα γίνει, θα γίνει σε εθελούσια βάση όπως οι συστάσεις. Ποια μορφή ε, θα πάρει ο τρόπος ε, υποβολής αιτήματο για να αξιοποιήσει κανείς αυτά τα κονδύλια. Αυτή η ερώτηση απευθύνεται προς όλους και είμαι ε, έτοιμος να ακούσω και να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ε, Κλείνοντα να επαναλάβω την έκκλησή μου να ε, δουλέψουμε γρήγορα, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό που σα είπα και περιμένω να ακούσω ε, του συναδέλφου και τι ενδιαφέρουσε ιδέες του. Το πιο σημαντικό όμω είναι ο προγραμματισμό ο ημερολογιακό για την έκθεση της τροπολογίας, την ψήφιση και ούτω καθεξή, για να μπορέσουμε να το κάνουμε μέσα στο 2016. Περιμένω και τα σχόλια των υπολείπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κρέλ, συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίω αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμά. Και κύριε Ντομπρόφσκι, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι χρειαστήκαμε κάποιο χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Δηλαδή ποιο είναι αρμόδιο γιατί. Και αυτό εξηγείται υπάρχει λόγος. Εξηγείται από το ότι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση έχει μια ασυνήθιστη δομή θα έλεγα. Γιατί αν δει κανείς ε, την πρόταση θα διαπιστώσει ότι η πρόταση αυτή εν μέρη εντάσσεται στην πολιτική συνοχή, δηλαδή είναι το κομμάτι εκείνο όπου στηρίζονται τα κράτη-μέλη για να προγραμματίζουν, να διαχειρίζονται και να υλοποιούν καλύτερα τα προγράμματά τους και νομίζω κατά το παρελθόν κάναμε πολύ καλή εμπειρία με την Task Force, παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα, η οποία Task Force ε, έδωσε τη δυνατότητα να εκταμιευτούν κονδύλια στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο. Και αυτό είναι αμφίβολα το κομμάτι το οποίο εντάσσεται στην πολιτική συνοχή. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος στην πρόταση της ε, Κομισιόν, το οποίο έχει άμεση σχέση με τα μακροοικονομικά. Έχει σχέση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με τεχνική αρρωγή και κανονικά όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πολιτική συνοχής. Αλλά και αυτά ε, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την τεχνική αρρωγή της ε, πολιτικής συνοχής. Και ρωτώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί τα κάνατε τόσο περίπλοκα. Γιατί στο κομμάτι που έχει σχέση με τις μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις όπου λέγεται ας πούμε ότι 60 εκατομμύρια από τα 120 εκατομμύρια αυτά είναι απαραίτητο να διατεθούν. Γιατί δεν βρήκατε στο ΕΚΟΦΗΝ κάποια αποθεματικά που είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσατε να έχετε βρει. Και γιατί τελικά δεν καταθέσατε ένα δικό σας πρόγραμμα. Γιατί κάνετε αυτή την περίεργη διασύνδεση μικρο και μακροοικονομίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Και το ερωτώ αυτό, διότι προφανώς ο κύριος Βανίστελ Ρόι και εγώ ε, διαπραγματευτήκαμε για τον γενικό κανονισμό και εσείς στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στις συστάσεις αναχώρα. Εμείς λοιπόν προσέξαμε, μεριμνήσαμε έτσι ώστε αυτά να μην ασκήσουν τη μεγάλη επιρροή που επιτιμούσαν οι Κομισιόν και το Συμβούλιο. Μεριμνήσαμε έτσι ώστε το πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής συνοχής να είναι απόφαση των κρατών μελών και όχι να λαμβάνονται αποφάσεις στο Συμβούλιο με βάση κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις χώρα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο προέκυψε και η αντιπαράθεση για τι ε, αρμοδιότητε. Κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε αποφύγει. Επανέρχομαι λιγάκι στο θέμα τη ε, χρηματοδότηση. Εδώ Πρόκειται για αύξηση του προϋπολογισμού για την τεχνική αρρωγή και αυτό έχει αυτό πάλι συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή στο συγκεκριμένο κανονισμό εμείς διαπραγματευτήκαμε να υπάρχει ένα εργαλείο όπου κράτη-μέλη τα οποία καλύπτουν κάποια προαπαιτούμενα και τα οποία επιθυμούν να στηρίξουν τη διοίκησή τους, αυτά τα κράτη-μέλη να μπορούν να απολάβουν την τεχνική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό, με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφώνεται η πολιτική συνοχής αποτελεσματικότερα. Αυτό λοιπόν το εργαλείο υπάρχει, μπορούν να κάνουν χρήση του εργαλείου και τα 28 κρατημέλη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε τον προϋπολογισμό για την τεχνική αρρωγή. Ερωτώ λοιπόν πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα αυτά δεν είναι δεσμευμένα, πώς ξαφνικά εμφανίζονται αδέσμευτα. Αυτά ήδη εντάσσονται στις υποχρώσεις και δεν καταλαβαίνω ε, πώς είναι δυνατόν να πρέπει να σκηθεί ειδική επιρροή έτσι ώστε να υπάρξει μεταφορά και από πλευράς ε, δημοσιονομικής ούτε και εδώ έχω καταλάβει πρέπει να σας πω πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μεταφορά γιατί κατά την άποψή μου στον κοινωτικό προπολογισμό δεν είναι δυνατόν δυνατόν να υπάρξει μεταφορά κονδυλίων ανάμεσα σε συγκεκριμένες γραμμές. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τους σκιώδεις εισηγητές από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη και Ατόματσικς. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντομπρόφσκης, αγαπητοί συνάδελφοι, Υποστηρίζω τις τροποποίησεις του κανονισμού, αυτό που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις στους διάφορους τομείς του δημοσίου. Ε, χρειάζεται πολύ συχνά χρόνος για να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να φανεί χρησιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Ε, γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν αρκετά νωρίς να ξεκινήσουν οι προσπάθειες. Δεν έχει σημασία τόσο μεγάλη αν πρόκειται για οικονομίες που έχουν πληγεί από την κρίση ή που είναι από την φύση τους αδύναμες οικονομίες. Δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή. Η καλύτερη πρακτική μπορεί να χρησιμεύσει σαν έμπνευση για εκείνους που θέλουν να ζητήσουν υποστήριξη. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι οι εταίροι, οι κοινωνικοί εταίροι, οι διάφοροι δημόσιοι φορείς να δεχτούν ο καθένας στο επίπεδό τους τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις και έτσι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί μεταξύ κρατών μελών και όλων των συμμετεχόντων εταίρων. Η βελτίωση της του περιφερειακού δυναμικού και του τοπικού δυναμικού πρέπει να είναι πτυχή κλειδί, πολύ βασική πτυχή, για κάθε προσπάθεια βελτίωσης του δημοσίων υπηρεσιών σε ένα κάτω μέλος στα πλαίσια της βελτίωσης του δυναμικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομείς ε, αρμοδιοτήτων. Πέραν αυτού θα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να δημιουργηθεί όμως αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε επίπεδο των κρατών μελών που θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Ο κύριος Μερζέ έχει το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, σίγουρα η τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη είναι κάτι το θετικό. Ωστόσο, δεν εγκρίνω και μάλιστα σε καμία περίπτωση την πρότασή σας σύμφωνα με την οποία θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα από τα κονδύλια της τεχνικής βοήθειας για τα, ε, ευρωπαϊκά, από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία και το ε, Ταμείο Επενδύσεων. Η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι κάτι με το οποίο είμαι κάθε τα αντίθετος και δεν καταλαβαίνω πώς δεν αντιτάσσεται η Επιτροπή Ρέτζη. Τα άρθρα 175 και 197 δεν επαρκούν στην τεκμηρίωση τη νομική του να, επιλεγεί αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης για την ε, συμμόρφωση με το ε, Σύμφωνο Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, ε, ε, στήριξης των διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων, εγείρει διάφορα ερωτήματα, γιατί έχετε διαλέξει πολύ συγκεκριμένους τομείς και θα ήθελα να τους υπενθυμίσω. Δικαστικός κλάδος, δικαστικό σύστημα, διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων, εκπαίδευση, αγορά εργασίας, συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας, κοινωνική προστασία, σύστημα δημόσιας υγείας, ε, πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κάνοντας αυτές τις επιλογές, ακριβώς αυτές τις επιλογές, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά παρουσιάζεται έναν οδικό πολιτικό χάρτη και ζητάτε από τα κράτη-μέλη να τον υπογράψουν. Και είναι οριστικά τρόπος παρέμβασης εισβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πάντοτε θέλει να προσανατολίζει τα κράτη παραπάνω από όσο θα ε, έπρεπε, όσο θέλει αυτή, προς μια απελευθέρωση ε, όλο και πιο έντονη και εντατική. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει καλύτερα εάν ήθελε ουσιαστικά να το παίζει ε, διαιτητής και διευθυντής των πάντων. Γιατί ε, αυτό δείχνει με τη στάση της. Έρχομαι τώρα στο θέμα της δημιουργίας π.χ. νέων ε, ε, ε, νέας φορολογίας, ε, επανεθνικοποίηση συγκεκριμένων πόρων, στόχος ενεργειακής αυτονομίας. Υπάρχουν και άλλες επιλογές πολιτικής και ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολήθηκε με αυτές. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι είδους στήριξη θα προσφέρει αυτό το πρόγραμμα στα κράτη-μέλη. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι τον ε, φίλο που πάντοτε όλοι έχουμε, ο οποίος βέβαια το καλό μας θέλει, αλλά τελικά με ένα περίεργο και στρεβλό ε, τρόπο ε, μας πλήττει. Ουσιαστικά με την πρόταση αυτή προσπαθείτε να μας φέρετε το δυστυχές, τη δυστυχή και θανάσιμη παρουσία της Τρόικας. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική βοήθεια που θα δώσετε στα κράτη-μέλη, που μπορεί να δοθεί από τα ε, κράτη-μέλη, δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι οι λαοί απορρίπτουν αυτές τις πολιτικές. Η βοήθεια, για παράδειγμα, που δίνεται στη Γαλλία για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας της δεν θα αλλάξει καθόλου τις κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή για την απόσυρση του νόμου ε, βάσει του οποίου ήδη εκατοντάδες ε, χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι και θα γίνει και στο μέλλον. Στην πρόταση αναφέρεται ότι μπορεί κανείς να στηριχθεί στους διεθνείς οργανισμούς. Θα ήθελα να ξέρω, για παράδειγμα, όταν μιλούμε για την αγορά εργασίας, θα κάνετε την επιλογή να βασιστείτε στις πρακτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ILO ή στις ε, πρακτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θέτοντας το ερώτημα αυτό, καταλαβαίνετε και την προτίμησή μου αλλά και τους φόβους μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ρέντ και η επόμενη σκιώδηση συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης που ήρθατε να συζητήσετε αυτή την πρόταση με εμάς. Νομίζω ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος. Μπορέσαμε να εξοικειωθούμε με αυτή, να προβληματιστούμε για να ξεκαθαρίσουμε τις ιδέες μας. Μιλάτε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζεται μια πολύ πολύχρωμη εικόνα της πραγματικότητας. Ε, τα παρουσιάζεται με ωραία χρώματα όλα και σαν να είναι πάρα πολύ καλά. Κάποιες από τις διαπιστωτικές μεταρρυθμίσεις είχαν καταστρεπτικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς στις διάφορες χώρες. Εξού και υπάρχει τόση υποψία για το τι ε, κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση, όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή, αλλά και σε πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρύτερα. Ναι, αυτή η πρόταση μπορεί να είναι ένα εργαλείο που θα δώσει δυνατότητες στα κρατη θα τα κάνει πιο ικανά να στηριχθούν στην τεχνική βοήθεια και στην εμπειρογνωμοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχή και να κάνουν μεταρρυθμίσει ευεργετικέ στις διάφορε χώρε. Όταν όμω βλέπουμε τον κατάλογο των θεμάτων που θέλετε να αντιμετωπίσετε, μπορεί τελικά από την πίσω πόρτα να θέλετε να εισάγετε μακροοικονομικέ πολιτικέ και να χρησιμοποιήσετε τα κονδύλια κοινωνική συνοχή για να πρόξετε πιο ψηλά στην ιεραρχία τη δική σας ή μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα ήθελα το θεματολόγιο αυτό να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ε, δουλέψουν χέρι με χέρι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεργαστούν για το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα κονδύλια για την οικονομική ανάπτυξη, για το καλό της κοινωνίας και να μην επιβάλλεται μια ατζέντα άνωθεν από τις Βρυξέλλες. Τά, το Ταμείο Συνοχής έχει επιτυχία όταν η προσέγγιση είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι εγκάρσια, οριζόντια και όχι από πάνω προς τα κάτω. Και θα πρέπει οι εθνικές αρχές βεβαίως να είναι, να είναι εμπλεκόμενες και να έχουν την ιδιοκτησία όλων αυτών των προτάσεων. Και τέλος. Μιλούμε για το ερώτημα των διαρθρωτικών ταμείων και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε εμείς στις περιφέρειες. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να στραφούν σε βιώσιμα project, σε βιώσιμα έργα, διότι μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους που αναφέρετε, θα δημιουργήσουμε απασχόληση και οικολογική αηφορία, βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τώρα η πρότασή σας πάει προς την άλλη πλευρά, δηλαδή να επιβληθεί η ατζέντα από τις Βρυξέλλες, τότε εμείς θα την αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ σκεπτικισμό και επιφυλάξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμάτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες δικές μου και επί της ουσίας και σε θέματα αρχής όσον αφορά το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, τέλη Νοεμβρίου η Κομισιόν πρότεινε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού και με βάση αυτά που γράφονται στο σκεπτικό η δημιουργία ενός κανονιστικού και θεσμικού υγιούς πλαισίου για την καλή λειτουργία της οικονομίας είναι καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, θέσεων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωση του επίπεδου ζωής και ε, βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά αυτά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ένα από τα βασικά αίτια για την χαμηλή απορροφητικότητα των διαρθρωτικών κονδυλίων οφείλεται τι ε, δυνατότητε που έχει η διοίκηση των κρατών μελών και η τοπική αυτοδιοίκηση. Από το 2014 στο 20 αυτόν τον προπολογισμό έχει υπάρξει ε, μια διασύνδεση ανάμεσα στην υγιή ε, διαχείριση και την πολιτική συνοχής η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσει την δική του την εταιρική σχέση για να μπορεί να, να στηρίξει τις συστάσεις που εκδίδει το Συμβούλιο. Ήδη στο τέλος του 2013 εισήχθη ένα στοιχείο το οποίο κατά τη δική μας άποψη το κίνημα των πέντε αστέρων έχει να κάνει και με την ίδια τη λογική τη ε, πολιτική συνοχή. Εμεί θεωρούμε ότι ο στόχο είναι να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στι διάφορε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να υπάρξει μεγαλύτερη ενταφική ακαιρότητα. Τώρα λοιπόν είμαστε συνομοθέτε και θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξη για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Πρώτα απ' όλα όμω, τι είναι αυτέ, ποιε εννοείται ακριβώ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, γιατί με βάση τον ορισμό στο site τη Κομισιόν υποτίθεται είναι μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική πρόνοια, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Και αν λιγάκι δούμε τι ακριβώς ε, σημαίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, σημαίνει ότι ε, χρηματοδοτούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, περικόπτοντας όμως κοινωνικά κονδύλια. Η πολιτική συνοχή, α μην ξεχνάμε, ότι σημαίνει κατ' ουσίαν 142 ε, εκατομμύρια ευρώ. Ε, θεωρώ ότι με βάση το άρθρο 23 η προσπάθεια να υπάρξει μια δική μας πολιτική συνοχή με μακροοικονομικά και μικροοικονομικά στοιχεία, αυτό πρέπει να έχει άμεση σχέση με τη συνοχή. Κατά την άποψή μου, και εδώ αναφέρομαι κυρίως στους συναδέλφους, ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να το ε, συσχετίζουμε με ένα πλωτικό πρόγραμμα μέχρι το 2020, γιατί υπάρχει ένα σκηνικό ε, του να ε, επηρεάσουν διάφορες μακροοικονομικές πραγματικότητες στον προπολογισμό και εκτός αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και διάφορα άλλα οικονομικά στοιχεία. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα τα εμπειρικά στοιχεία, αυτά να τεκμηριωθούν, γιατί όλα αυτά είναι εις βάρος των επιδοτήσεων. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο δύσκολο να μιλάμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αυτός που είναι ο στόχος ε, σε τελική ανάλυση είναι ακριβώς να αναθεωρηθεί η πολιτική συνοχής, όχι όμως να στρεβλωθεί. Και είναι αλήθεια ότι το κράτος μέλος μόνο του θα αποφασίσει αν θα ζητήσει βοήθεια για το πρόγραμμα. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά πότε και πώς ε, οι πιο αδύναμες χώρες ε, ε, επηρεάζονται από τις αναχώρασεις συστάσεις. Και ποιος δεν θέλει να βελτιώσει τη γραφειοκρατία, τη δικαιοσύνη, την φοροδιαφυγή. Στη δική μας την περίπτωση εμείς ζητήσαμε επανειλημμένα και σε κείμενα που έχουν ψηφίσει στην Ολομέλεια την ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων των περιφερειακών και τοπικών αρχών όλα αυτά έχουν ένα στόχο, δηλαδή την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, κατ' ουσίαν τι σημαίνουν, σημαίνουν ή περικοπή των ε, συντάξεων και άλλων κοινωνικών ε, παρεμβάσεων. Και αν γίνουν όλα αυτά, δεν καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν επιπτώσει στη ζωή των πολιτών. Γι' αυτό γελάω με πικρία. Ε, την Ελλάδα, την αναφέρατε ως παράδειγμα για την Τρόικα η ε, ανεργία των νέων έχει φτάσει μέχρι και το 50% και έχουμε ένα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ε, που έχασαν την εργασία τους ε, και πάνω από 2 εκατομμύρια Ελλήνων που έχουν χάσει την υγειονομική περίθαλψη το μάντρα των διαρθρωτικών δεθμίσεων, όπως επίσης και η ε, πολιτική λιτότητα. Σε αυτά για μας είναι άχρηστα αλλά και επικίνδυνα. Επίτροπε, συνάδελφοι, είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει ένα περαιτέρω στοιχείο το οποίο για άλλη μια φορά υποτίθεται θα στηρίξει την πολιτική συνοχή. Μα είναι αλήθεια αυτό. Thank you, thank you, Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Σαν σκιώδη εισηγητή εκ μέρου των φιλελευθέρων, δεν έχουμε παρόντα τον σκιώδη εισηγητή τη Άλντα και είμαι ο μόνο εκπρόσωπο τη Άλντα εδώ. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τη θέση μα σαν ομάδα τη Άλντα. Σύντομα. Να τονίσω δύο πράγματα. Ήδη έχουμε τη μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής. Μία από τις απαιτήσει της νέας μεταρρυθμισμένης πολιτικής συνοχής είναι ο κατάλογος αιρεσιμοτήτων που ανήκει στις διάφορες εταιρικέ συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι αιρεσιμότητες στις περισσότερες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν απαιτήσει για διαθωτικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε το προτινόμενο πρόγραμμα σχετίζεται στενά με τα προβλήματα της πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, υποστηρίξαμε τις ζυμώσεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δύο φορές το χρόνο θα έχουμε συστάσεις αναχώρα. Και αυτό το υποστηρίζουμε και συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Αυτό σχετίζεται με τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάποια κράτη-μέλη γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που απαιτείται για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν όμως κράτη-μέλη στα οποία απαιτούνται διαθωτικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται για να υποστηρίξουν την εφαρμογή των πολιτικών συνοχής. Παράδειγμα, για ένα κράτος μέλος. Τη δική μου χώρα. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουν στόχο να υποστηρίξουν τις υποδομές υγείας για τις υπηρεσίες αυτές. Όμως, η μεταρρυθμίση του τομέα της υγείας δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι δυνατόν να στείλουμε υποστήριξη από τα διαθωτικά ταμεία, διαθωτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαθωτική μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας της Βουλγαρίας. Χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη. Χρειαζόμαστε αυτού του είδους τη βοήθεια. Και εδώ είναι το προσωπικό μου ερώτημα. Συνήθως θεωρούμε ότι αυτού του είδους υποστήριξη θα πρέπει να προέρχεται από την τεχνική αρρωγή των διαστατικών ταμείων. Από τεχνική αρρωγή η οποία ήδη έχει προγραμματιστεί μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ τεχνικής αρρωγής και του νέου προγράμματος και πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που θα υποστηρίζονται από αυτές τις δύο πτέρυγες από τα ίδια διεθνωτικά ταμεία, διότι μιλάμε για διεθνωτικά ταμεία. Το νέο εργαλείο στα πλαίσια των διεθωτικών ταμείων. Αυτή είναι η θέση και η ερώτηση που έχω να εκφράσω εκ μέρους της ΑΛΔΕ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να δώσω το λόγο τώρα στον φιλοξενούμενό μας, τον εισηγητή από την Επιτροπή Γεωργίας, όχι, α, απασχόλησης, με συγχωρείτε, συγγνώμη, από την Επιτροπή Απασχόλησης, τον κύριο Σόγκαρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η Επιτροπή Απασχόληση θα, θα είναι στη διαπραγματεύση στη θέση 53 συν οι επιτροπές μας όμως θα συνεργαστούν άριστα πιστεύω. Είναι σημαντικότατο το νομοθέτημα. Και πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τα θέματα της απασχόλησης, όπως τους αξίζει. Έχουμε χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, έχουμε υψηλή ανεργία και είναι ανησυχητική η ανεργία των νέων που είναι μακροχρόνια. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστέ διευθυντικέ μεταρρυθμίσεις για να προωθήσουμε τι επενδύσει, να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα την οικονομική και να αναπτύξουμε τι αγορέ Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα από ποτέ. Συμφωνώ με, την, με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάζεται λιγότερο εξωθετήσεως νέων νομοθετημάτων, αλλά καλύτερα ανταυτού να εφαρμόζει αποτελεσματικότερα τα ήδη φυστάμενα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων. Ένα από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η καταχώρα συστάσεις. Το χαμηλό επίπεδο εφαρμογή των μέτρων σε διάφορα κάτι μέλη κυρίως στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών είναι εμπόδια για την ανάπτυξη και για ένα περιβάλλον που είναι φιλικό για τις επενδύσεις και για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό η δημιουργία ενός μόνιμου προγράμματος υποστήριξης εθνωτικών μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένο προπολογισμό έχει μέγιστη σημασία. Τέτοια υποστήριξη, αν ήταν διαθέσιμη στη χώρα μου, τη Ρουμανία, πιστεύω ότι το ποσοστό απορρόφησης στην περίοδο 2007-2013, σε αυτή την προγραμματική περίοδο, δεν θα ήταν μόνο 70% και δεν θα βλέπαμε τις καθυστερήσεις στο σχεδιασμό επιχειρησιακών προγραμμάτων εν μέρη που οφείλονται συνέλευση στατηγικών σε ζωτικού τομεί. Η τεχνική υποστήριξη δεν θα πρέπει να είναι μόνο διαθέσιμη σε περίοδο κρίσεων. Είναι καλύτερο να απολαμβάνουμε νέα χρήση νέα κρίση συγγνώμη, και να δημιουργούμε ανθεκτικές οικονομίες οι οποίες να μπορούν να αντέξουν σε μελλοντικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλμπρεχτ, εκ μέρους Επιτροπής Υπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί και τι κάνει το Κοινοβούλιο και δεν περιμένετε πιστεύω ότι θα εργαστούμε χωρίς ενδελεχέστερη ανάλυση. Περί τίνος πρόκειται. Είδαμε ερωτήσει που ετέθησαν, που δείχνουν ότι δεν είναι τα πάντα σαφή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διευκρινήσει. Θα ακολουθήσω την Κωνσταντς και τον Λάμπερτ με την ερώτηση. Πρέπει να καταλάβουμε πώς σκέφτεστε, αν έχουμε τις συστάσεις κατά χώρα. Οι χώρες πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις. Αν προτείνεται ένα νέο εργαλείο, τι σημαίνει αυτό. Ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά ή αυτό που λείπει είναι τα χρήματα. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, δεν έχουμε μεγάλα ποσά. Τα χρήματα που θα είναι κίνητρο για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο, αυτό καταλαβαίνω. Σας προτείνουμε ένα εργαλείο για να το ενστερνιστείτε και να κάνετε τη μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα όμως λέτε ότι αυτό είναι επιθελοντικής βάσος. Αν θέλετε να κάνετε τη μεταρρύθμιση, μπορείτε να στηριχτείτε από μας. Αλλά δεν θέλετε να πάρετε την υποστήριξή μας. Σημαίνει ότι δεν θα κάνετε μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η πρόταση, όπως καταλαβαίνω. Σας προσφέρουμε το εργαλείο. Για να δουλέψετε καλύτερα. Ένα κίνητρο δηλαδή. Σας προτείνουμε να το κάνετε. Διότι δεν το κάνετε. Γι' αυτό σας προτείνουμε το εργαλείο. Αν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αν τα κάτι μελη κάνουν τις μεταρρυθμίσεις... δεν χρειαζόμαστε το εργαλείο. Ωραία. Ερώτηση. Προτείνουμε το εργαλείο, το οποίο το πήραμε από συγκεκριμένο κομμάτι του προπολογισμού. Αν το παίρνουμε από συγκεκριμένο σημείο του προπολογισμού υπάρχουν συνέπειε. Το ερώτημα του Λάμπερτ ήταν, ποιο θα το κάνει. Αν πάρουμε τα χρήματα από τα ταμεία, δεν σημαίνει ότι αυτά θα πάνε στην περιφερειακή ανάπτυξη, DG Radio κλπ. για την πολιτική συνοχής. Αν είναι περί πολιτικής συνοχής και συζητούμε αυτό το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που συνδέεται άμεσα με την πολιτική συνοχής, διότι οι συστάσεις κατά χώρα δεν αφορούν την πολιτική συνοχής μόνο. Αυτά τα χρήματα θα πάνε λοιπόν σε κάτι σχετικό με την πολιτική συνοχής. Δεν σημαίνει ότι τα χειρίζεται η DG Regio. Δεν τυχαίο ότι στο Κοινοβούλιο, εδώ έχουμε την Επιτροπή την Περιφερειακή που το εξετάζει. Σημαίνει ότι είναι πρόβλημα συνοχής. Ερώτηση, ποιος θα το αναλάβει και πώς θα το εφαρμόσει. Και άλλη ερώτηση, που είναι ερώτηση που ακούτε στην αίθουσα. Ωραία. Αν τα κράτη-μέλη μας πούν ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη, καλώς. Έχετε τα χρήματα, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά προτείνετε ένα σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει θα πάρετε χρήματα, αλλά θα σα προτείνουμε του εμπειρογνώμονε. Θα σα προτείνουμε εμεί το Διεθνή Οργανισμό. αυτή είναι η απειλή, ο φόβο. Αυτό έχετε υπόψη σα. Συγκεκριμένου φορεί που μπορούν να βοηθήσουν συγκεκριμένε χώρες να κάνουν αυτό που πρέπει. Ποιο αποφασίζει ποιο θα επιλεγεί. Διότι υπάρχει ένα μενού στην πρότασή σας. Αυτός που προτείνει κάνει πολιτική επιλογή. Γι' αυτό κάποιοι συνάδελφοι φοβούνται ότι θα προτείνετε συγκεκριμένους φορεί που θα προτείνουν συγκεκριμένη πολιτική. Άρα αυτό είναι ένα κρυμμένο στοιχείο που προωθεί συγκεκριμένη πολιτική. Λοιπόν, Επίτροπε, αν έχετε την καλοσύνη να μα πείτε, να διευκρινίσετε, ίσως όχι σήμερα, ξεκαθαρίστε τα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Ποια είναι η λογική όλου αυτού, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, πηγαίνει σύμφωνα με την πολιτική συνοχή. Τρίτον, πώ θα λειτουργήσει αυτό, ποιο αποφασίζει ποιο θα βοηθηθεί και ποιο θα βοηθήσει, διεθνή οργανισμό, εμπειρογνώμονε κλπ. Τα κράτη-μέλη θα έρθουν πρόταση και εσεί θα πείτε όχι, αυτό, το άλλο όχι, το άλλο ναι. Δεν σας δίνουμε χρήματα, άρα εμείς αποφασίζουμε ο ποιος θα πληρώνεται. Ή υπάρχει ελευθερία επιλογής. Πολιτικός πώς αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις από τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και τους προσκεκλημένους εισηγητές άλλων επιτροπών. Επιτροπέ, ε, έχετε το λόγο πριν ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Παρακαλώ. Βεβαίως και θα έχουμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αρκετά τα ερωτήματα. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να το ομαδοποιήσω και να απαντήσω συνολικά. Ως προς τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Όπως ήδη είπα, στην εισαγωγική μου παρέμβαση και όπως φαίνεται στην πρόταση, τα χρήματα προέρχονται από την τεχνική βοήθεια, η οποία γίνεται αντικείμενο κεντρικής διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παίρνει 112,2 εκατομμύρια από το ΕΣΥΦ και 30,6 από το ΕΤΠΑ. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτά είναι τα χρήματα της τεχνικής βοήθειας που διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, τίθεται το ερώτημα, θα υπονομεύσει αυτό την ε, δουλειά της τεχνικής βοήθειας. Εγώ σας είπα ότι πράγματι έχουμε υψηλότερα ποσά στην τεχνική βοήθεια σε αυτή την προγραμματική περίοδο συγκριτικά με τις προηγούμενες. Έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα στην τεχνική βοήθεια από ό,τι πριν. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί και αξιολογεί ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες και της τεχνικής βοήθειας και του ε, νέου προγράμματος της πρότασης που προτείνουμε. Τώρα, το ερώτημα, εάν τα χρήματα αυτά αφορούν το σύνολο της περίοδου, η απάντηση είναι ναι. Για την αναδιοργάνωση του επιτελείου, του προσωπικού. Να σας πω ότι είναι μια υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίσει αυτή τη δουλειά. Αναφέρθηκε η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ δεν ασχολείται όμως αυτή. Είναι η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διοικητικά υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρεται κατά βάση στον πρόεδρο Γιούνκερ και σε μένα. Και συντονίζει αυτή η υπηρεσία όλο αυτό το έργο ε, σε σχέση με τις λοιπές γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εξωτερικούς φορείς παράγοντες εμπειρογνώμονες εάν αυτό χρειάζεται. Αυτά για τη διοικητική της υπόσταση. Δεν ανήκει δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ, είναι ξεχωριστή υπηρεσία. Τώρα, κατά πόσο θα επιβληθεί στα κράτη-μέλη να κάνουν το ένα ή το άλλο πράγμα. Θα ήθελα να επαναλάβω το εξής είναι εθελούσια ε, η, υπαγωγή σε αυτό το πρόγραμμα και εξαρτάται από το αίτημα. Το κράτος μέλος πρέπει να αιτηθεί τεχνική βοήθεια. Τώρα ποιος θα αποφασίσει τα πώς και τα γιατί να σας πω ότι γίνεται αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δεν θα επιβληθούν ούτε οργανώσεις, ούτε φορείς, ούτε εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα προκύψει κατόπιν αιτήματο του κράτους μέλους. Τώρα, για τη σχέση με την πολιτική συνοχής το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ποια σχέση έχει με την πολιτική συνοχή. Απαντώ λέγοντας ότι πράγματι αυτό έχει συζητηθεί εκτεταμένα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι η υπηρεσία στήριξης με διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ε, συνεχίζει το έργο της Task Force για την Ελλάδα και της ομάδας στήριξης της Κύπρου Και αν πάρουμε το παράδειγμα της Task Force για την Ελλάδα, η υπηρεσία αυτή βοήθησε έτσι ώστε να βελτιωθεί δραματικά η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα. Βεβαίως λήφθηκαν εξωτερικές αποφάσεις για διευκόλυνση των χρηματικών και ταμιακών ροών, όμως η Tax Force για την Ελλάδα ε, κόμισε τεχνική βοήθεια για την ευελτίωση ε, της χρηματοδοτικής ροής και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τέτοιου είδου τεχνική βοήθεια είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη μόνο για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Τώρα όμως μιλούμε για μια υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που μπορεί να προσφέρει τεχνική βοήθεια και σε χώρες που δεν βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής κατόπιν αιτήματό του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την εξή αξιολόγηση και εκτίμηση. Θεωρεί ότι με την ε, τεχνική αυτή βοήθεια μπορούμε να εντοπίσουμε και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνέργειες. Να βάλουμε μαζί την εθνική χρηματοδότηση με το ευρωπαϊκό κονδύλια, να δούμε την ατζέντα και το θεματολόγιο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναλόγως με το πώς το ζητά το εκάστοτε κράτος μέλος. Πολλοί είπαν το εξή. από εδώ έχουμε τεχνική βοήθεια, από εκεί έχουμε ε, κονδυλία για τη συνοχή και να μην υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι είναι καλό να, ξεπεράσουμε αυτό το τείχος και να δούμε εκεί που μπορεί να υπάρχουν συνέργειες, συνέργειες και γι' αυτό έχουμε μια δομή που συντονίζει τις διάφορες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρει συνέργειες μεταξύ όλων αυτών των δράσεων και κάποια παραδείγματα που πρόβαλε η κυρία Πρόεδρος είναι ακριβώς τα παραδείγματα που αναδεικνύουν ε, το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή η τεχνική βοήθεια. Τέθηκε το εξή ερώτημα. Μήπως είναι άλλη μια απόπειρα η πολιτική συνοχής να υποταχθεί στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πω ξεκάθαρα όχι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Και συμφωνώ με τις απόψεις ορισμένων συναδέλφων. Έχουμε τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις, έχουμε τον κανονισμό για τα διάφορα ταμεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, τα κοινωνικά θέματα, η, πολιτική, η κοινωνική πολιτική. Είναι παιδεία στα οποία δραστηριοποιούνται αυτά τα ταμεία και θα πρέπει, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές προκλήσεις. Την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα κοινωνικά προβλήματα. δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα αλλάξουμε αυτά. Είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Υπάρχει προγραμματική περίοδος 7 ετής και δεν θα υπάρξει επαναπρογραμματισμός. Κάθε ειδική σύσταση αναχώρα θα προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Επομένως, το θέμα είναι κατά πόσο σε ορισμένες συνθήκες οι μεταρρυθμίσεις που που μπορεί να βρίσκονται ή μπορεί και να μην βρίσκονται στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποστηριχθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι αυτή η προϋπόθεση για να μπορέσουν οι χώρες να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκά κονδύλια. Και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η τεχνική βοήθεια μπορεί να αξιοποιηθεί για να ε, συνδεθεί τι το, συνδεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αυτές τις πολιτικές. Εμείς πιστεύουμε ότι τελικά θα γίνει πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο εκάστοτε κράτος μέλος. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό απαντώ στο ερώτημά σας, για το γιατί η πρόταση αυτή είναι ευρεία. Πράγματι είναι μια ευρεία πρόταση, εσκεμένα, γιατί θέλουμε να περιλάβουμε όλες τις δυνατότητες, θέλουμε να μπορούμε να λειτουργήσουμε πάνω σε διάφορους και διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Τα κράτη-μέλη ζητούν βοήθεια για ορισμένους τομείς ε, πολιτικής και μπορούν να εξετάσουν πώς τα διαθέσιμα εργαλεία για άλλες πολιτικές μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Βεβαίως μπορεί να συμφωνήσουμε πάνω σε έναν ακριβή κατάλογο ή και όχι. Και βεβαίως θα συζητηθούν όλα αυτά τα πεδία. Δράσεις. Αλλά πάντοτε το κράτος μέλος θα το ζητά αυτό και θα θεωρεί ότι είναι αυτό παρέντητο για να καλύψει τις ε, δικές του ανάγκες. Και τώρα, ποιοι διεθνείς ε, φορείς θα εμπλακούν. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο εξαρτάται από την περίπτωση. Όταν συζητούσαμε τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με την ελληνική κυβέρνηση. Είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση ερωτήσεις για ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που είχαν ε, εφαρμοστεί και είχε πάρει την απάντηση ότι η εμπειρογνωμοσύνη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θα αξιοποιηθεί. Ο ILO δηλαδή θα εξετάσει τις προτάσεις μεταρρύθμισης και θα υποβληθεί πρόταση αναλόγως. Επομένως, οι διεθνείς οργανισμοί ε, μπορεί να διαφέρουν αναλόγως με την περίπτωση. Τέθηκε το εξής ερώτημα. Για τη χαμηλή απορροφητικότητα η οποία συχνά συνδέεται με τη χαμηλή διοικητική ικανότητα και αυτό αληθεύει συχνά και πιστεύουμε εμείς ότι η πρόταση αυτή επιλύει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Αναφερθήκατε και στην απλούστευση η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την πρόταση αυτή, το παραδέχομαι, όμως η απλώστευση αποτελεί μέρημνα και μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα υποβάλει πρόταση για την απλούστευση ε, του συστήματος διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Ταμείων και Κονδυλίων των διαφόρων μέσα σε αυτά τα ταμεία και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτης ελπίζουμε ότι θα μας στηρίξει στην πρότασή μας αυτή. Πολύ συχνά εμείς υποβάλλουμε προτάσεις απλούστευσης και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έρχονται και επιβάλλουν επιπρόσθετες στιβάδες, στρώματα ελέγχου ε, για να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς. σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την απλούστευση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτά προς το παρόν νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα πεδία, τις περισσότερες ερωτήσεις. Περιμένω με ενδιαφέρον το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Δύο ονόματα, δύο, δύο ονόματα έχω στον κατάλογό μου. Μαλέτιτς. Thank uh, Σας καλωσορίζουμε, κύριε Ντομπρόφσκης. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με όλους τους ε, συναδέλφους ε, που είπαν ότι το πρόγραμμα αυτό, SRSP, είναι βεβαίως και πρόσδεκτο για καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Έχω όμως ε, κάποιες ερωτήσεις. Η μία ερώτηση έχει σχέση με αυτό που υπογράμμισε η κυρία Μιχαήλοβα. Ε, νομίζω ότι ε, δεν τοποθετηθήκατε ακριβώς ε, σε αυτή την ερώτηση και χρειαζόμαστε κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι προφανώς ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα ε, με όλους τους άλλους ε, παράγοντες. Ε, είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με την Task Force σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων για θέματα τεχνικής αρρωγής. Αλλά κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το πώς ε, μπορούμε να προσεγγίσουμε συγκεκριμένα κάποιες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρες έχουμε επιχειρησιακά ε, προγράμματα σε εθνικό, σε άλλα σε περιφερειακό επίπεδο και η τεχνική βοήθεια αφορά διαφορετικά προβλήματα τα οποία και αυτά έχουν σχέση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συντονίζουμε την συμπληρωματικότητα σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό είναι το ένα ερώτημά Το άλλο έχει σχέση με το μέλλον του υποστηρικτικού προγράμματος. Διαπίστωσα ότι προβλέπεται ενδιάμεση αξιολόγηση ε, στα μέσα του 2019. Αλλά τότε είναι πολύ αργά. Ε, για να σκεφτεί κανείς ε, το μέλλον των ε, προγραμμάτων πολιτών, δημοσιονομικών προγραμμάτων. Εσείς μήπως έχετε κάτι άλλο κατά νου για το μέλλον, πέρα από την ή μετά την περίοδο του 2019-20. Και το τρίτο ερώτημά μου είναι κατά πόσον υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και του γεγονότος ότι θα εφαρμόσετε μακροοικονομική αιρεσιμότητα σε μία περίπτωση, αλλά στην περίπτωση όπου η χώρα αυτή δεν καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν θα ζητήσει και βοήθεια. Γιατί είπατε ότι όλα αυτά εξαρτώνται και από τη ζήτηση. Πιστεύετε πραγματικά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να στραφώ σε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ε, τέθησαν. Οι συστάσεις κατά χώρα έχουν ολοκληρωθεί και προσανατολίζουν τη δράση των χωρών προς στόχους μακροοικονομικούς που δεν σχετίζονται με τους μικροοικονομικούς στόχους, μακροοικονομικούς λοιπόν στόχους οι οποίοι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να επιτευχθούν, διότι είναι συγκυριακές πολιτικές αυτές. Και πρέπει να επαναπροσανατολιστούν οι, οικονομι... οι οικονομίες της Ευρώπης προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν και διαθετικά στοιχεία που αναφέρονται όλο και περισσότερο και αφορούν στοιχεία μεγάλης κλίμακας, εθνικής κλίμακας και μακροοικονομικού είδους. Λοιπόν, κάποια πράγματα που λέτε και αναφέρετε στον κατάλογο υπάρχουν. Μετά, η, η απόφαση, η κρίση, κατά πόσο, οι συστάσεις, η τεχνική αρρωγή που θα χορηγηθεί αρκεί, είναι αρκετά ευέλικτη για να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι των διαφόρων χωρών. Αυτή είναι μια άλλη κρίση, μια άλλη απόφαση που προσωπικά επιφυλάσσομαι να αποφασίσω. Διότι δεν υπάρχει πολιτική ευθυγράμμιση όλων των χωρών. Στην επιδίωξη διαθωτικών στόχων υπάρχει ελευθερία για διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Διότι είμαστε ενωμένοι στην διαφορετικότητα και όχι στην ισότητα. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μας σήμα, αν θέλετε, που προβάλλουμε. Κάποια πράγματα εδώ μέσα όμως έχουν χαρακτήρα περισσότερο μικροοικονομικό, όπως η γεωργική πολιτική, η αγροτική πολιτική είναι πολιτική τομεακή που προσπαθεί να καταστήσει αποτελεσματικές και παραγωγικές τις γεωργικές επιχειρήσεις και έχει μια λογική που διέπεται από κατά περίπτωση ε, πολιτική, επιτροπές κατά περίπτωση κλπ η διαθροτική πολιτική, η πολιτική της συνοχής, η περιφερειακή πολιτική, όπως το ονομάσουμε και κοινωνική που σχετίζεται με το κοινωνικό ταμείο ή αφορά μικροοικονομικές πολιτικές που χρειάζονται χρόνο. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο και δημιουργούν πιο αποτελεσματικά συστήματα οικονομικά στον τομέα των υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα κλπ. Για το Ταμείο Αναπτύξης Υπέθρου μιλάμε για την Γεωργία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γεωργικό τομέα που συνδέεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο με την υπόλοιπη οικονομία. Έχουμε πολιτικές πολύ διαφορετικές και κάθε μια πολιτική έχει τα εργαλεία της, τα ειδικά, την τεχνική της αρρωγή, τη δυνατότητα προσανατολισμού των δράσεων, όχι τόσο των χωρών, αλλά των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα, τις διάφορες επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε όμως να είμαστε προσαρμοσμένοι εδώ στις τάσεις κατά χώρα που εδώ μιλάμε για ε, γενικές πολιτικές μακροοικονομικού είδους. Εδώ βλέπω έναν κίνδυνο μεγάλης σύγχυσης μεταξύ των δύο. Προσωπικά λοιπόν, πέρα από τις κρίσεις και αποφάσεις και κρίσεις που θα εκφράσει κάθε πολιτική ομάδα, χρειάζεται ένας προβληματισμός. Στο κατά πόσο τον κατάλογο πρέπει να βγάλουμε από εδώ θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις μεγάλες διαθρωτικές γενικές πολιτικές. Αντιθέτως σχετίζονται με τομεακές πολιτικές που έχουν μια λογική δική τους και δικό τους χρόνο υλοποίησεως πολιτικές για εις βάθος μεταρρύθμιση της οικονομίας της χώρας. Γι' αυτό μιλάμε για διαθωτικές αλλαγές και πολιτικές. Χρειάζονται χρόνο, υπομονή, ικανότητα, αρμοδιότητες πολύ ειδικέ. Κάτι που δεν θα μπορούν να έχουν οι δικοί σας ειδικοί. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εισβολής, αν θέλετε, άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά κάποια πράγματα δεν βρίσκονται στην παρουσίαση που κάνατε. Ούτε και στα θέματα που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Εάν δεν ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση, κάποιος ε, θα θεωρούσε ότι είναι μια επέκταση της Τρόικας επιθελοντικής βάσης. Θα γίνει αντιληπτή η προσπάθεια αυτή σαν μια εισβολή ε, ε, από πλευράς διαφόρων τομέων που με μεγάλη ικανότητα διάφοροι τομείς και με διάφορους περίπλοκους μηχανισμούς αντιμετωπίζουν τις πολιτικές ε, της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όλες θα ήταν καλά. Δεν είναι αυτός ο στόχος ούτε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ούτε και στις τάσεις κατά χώρα που θα αποτελούν πλέον πλεονασμό και δεν θα ακολουθούνται. Είναι λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς από τον ένα χρόνο στον όλο. Και κυρίως εδώ δεν υπάρχει γεωργική πολιτική, δημόσια υγεία δεν συμπεριλαμβάνεται, δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταρρύθμιση της βοήθειας στον τομέα της υγείας. Το να προτείνεται μια μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα πρέπει να εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορά θέματα οικονομικά και χρηματοστατικά, διότι εδώ έχουμε άλλη πολιτική λογική στη τομή. Η μεταρρύθμιση κοινωνική δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα οικονομίας ή πολιτικής της υγείας. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, το οποίο απαιτεί άλλο χρόνο και άλλου είδους ε, τεχνική αρρωγή. Ευχαριστώ κύριε Σπυράκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ε, κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν στην τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα. Όπως ε, γνωρίζετε πολύ καλά, στο, στην ανακοίνωση του Eurogroup ε, υπάρχει δέσμευση να χορηγηθεί τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να προαχθεί ανάπτυξη. Και με βάση την έκθεση Υπουργείου Οικονομικών που πρόσφατα κατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν υπάρχει ικανοποιητική απορροφητικότητα. Όπως μας, είπε, μας είπατε, η τεχνική βοήθεια είναι μετά από έτοιμα. και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η Task Force ε, στην πρώτη της ε, θητεία δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή για την Ελλάδα και επίσης θα υπάρξουν κάποιες άλλες λύσεις ε, που να προταθούν από την Ελλάδα θα προταθούν από κάπου αλλού για να υλοποιηθούν οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις τις οποίες έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ε, συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η κυρία Μπρέσσαου. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η πρόταση ως έχει κατατεθεί είναι θετική. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρώσουμε ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά την ανώριμη επιλογή μέτρων για την οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα και όχι απαραίτητα μόνο στις ε, οικονομικά αντίναμες χώρες. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη νομοθετική ε, εφαρμογή, εφαρμογή των νόμων σε όλα τα κράτη-μέλη. Οφείλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με το ποια θα πρέπει να είναι η σωστή χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Και να δούμε λιγάκι τα κονδύλια που έρχονται από τα ε, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και από, τα, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε με την ε, οικονομική πολιτική και την πολιτική συνοχή, που κατ' ουσίαν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα δηλαδή πρέπει να προσέξουμε. Και θέλω να πω το εξής. Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν δικούς τους ε, στόχους, και αυτές, ε, αυτοί οι στόχοι αναφέρονται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος, ένας στόχος πολιτικής συνοχής είναι η υποστήριξη της οικονομικής και εδαφικής ε, συνεργασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως ε, μέσα από την στήριξη των επενδύσεων, την βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Η υποστήριξη των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καταρχήν δεν έχει πολλά ε, κοινά στοιχεία με την πολιτική συνοχή, αλλά έχει κοινά στοιχεία με τη χρηματοδότηση. Ο κ. Ζωμαζουέ και η κυρία Κρέλ τα ανέφεραν αυτά. Και διαρωτώ με κατά πόσον η Κομισιόν μπορεί να αναφερθεί συγκεκριμένα στις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος. Και όσον αφορά και τον τομέα υπαριθμών 5 του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό αναφέρομαι κυρίως. Και θέλω να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Νομίζω ότι ο κατάλογος των ε, προσυποστήριξης ετοιμάτων από το πρόγραμμα προφανώς και πώς θα εγκρίνονται τα αιτήματα αυτά και η εφαρμογή της ε, των νομοθετικών ρυθμίσεων που προκύπτουν, αυτά είναι καθοριστική σημασία. Αναφέρθηκαν και από άλλο συνάδελφο. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε τις προτάσεις από αυτό το πρόγραμμα να τις εντάξουμε περισσότερο στις εταιρικέ ε, συμφωνίες. Εκεί πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Βεβαίως ε, αυτό είναι ε, προκαλεί χρόνο τριβή αλλά το θέμα είναι πόσο συμπληρωματικά είναι όλα αυτά. Και τέλος, όσον αφορά την επικάλυψη των εργασιών και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων. Και εδώ αναφέρομαι κυρίως στα προγράμματα, στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020. Ο κύριος Ζέλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ έριξα μια ματιά μόνο σε αυτό το έγγραφο, δεν είχα άλλο περιθώριο, αλλά να σας πω το εξή. Κοιτάξτε, εγώ αποκόμισα την εντύπωση ότι πρόκειτο για τεχνική βοήθεια και ότι θα μιλήσουμε για διαρθρωτικά ταμεία και για την πολιτική συνοχή. Αυτό θα το κάνουμε για να δώσουμε ένα εργαλείο στα κράτη-μέλη έτσι ώστε η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και των επιχειρησιακών προγραμμάτων αυτή η καθυστέρηση να αρθεί, να ξεπεραστεί. Αυτό Αναφέρεται επανειλημμένα ότι υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν το διοικητικό δυναμικό είτε γιατί δεν είναι σωστά και επαρκώς εκπαιδευμένοι οι συνεργάτες είτε γιατί δεν επαρκεί το προσωπικό για να εφαρμοστούν αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Διάβασα όμως τελικά και την πρόταση κανονισμού και ξέρετε κάτι, κατέληξα σε τελείως διαφορετική εντύπωση. Δηλαδή κατ' ουσίαν πρόκειται για ορισμένες χώρες όπου έχουν υπάρξει μεταρρυθμίσεις, παρόλα αυτά όμως δεν παρουσιάζουν οικονομική ανάπτυξη παρά τις μεταρρυθμίσεις και το θέμα είναι να τους δώσουμε μια καλή διακυβέρνηση, good governance. Σήμερα και με την πολιτική διεύρυνσης μπορέσαμε σε ορισμένα κράτη και πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους διαθέσουμε κάποιες δυνατότητες για να βελτιώσουν τη διοίκησή τους, να μπορούν να εφαρμόζουν καλύτερα τις την κοινοτική νομοθεσία. Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Ελλάδας από κάποιους. Όπου σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα στείλαμε Task Force. Και γιατί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει κάποιες προτάσεις που έχουν και σχέση με την κυριαρχία ενός κράτους, κάτι όμως που δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το στείλαμε. Και έτσι κρίνουμε ότι το συγκεκριμένο κράτος μπορεί στο μέλλον να ενταχθεί καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και μέχρι εδώ καλά. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι κάποια κράτη που έχουν ε, δυσκολίες θα πρέπει να βοηθηθούν. Ε, αναφέρθηκε συγκεκριμένα το άρθρο 8 και όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν οι οποίε όμω αυτέ δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με την πολιτική συνοχή. Αφορούν όμω όλα αυτά ε, τον τρόπο διακυβέρνηση μια χώρα και υποτίθεται εμεί θέλουμε να βοηθήσουμε. Είδα λιγάκι του αριθμού 142 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η αριθμή. Και διερωτώ με, τι δυναμικό μπορούμε να διαθέσουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα διαθέτουμε 35 εκατομμύρια αν υπολογίσουμε το κόστος ενός εμπειρογνώμονα 100.000 το χρόνο, χαμηλό μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαθέσουμε 350 εμπειρογνώμονες ανά έτος, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Για μένα σημαίνει αυτό ότι τα κλασικά επιχειρησιακά προγράμματα δεν μπορεί να εννοούμε αυτά, γιατί από τα 28 κράτη-μέλη έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρησιακά προγράμματα που διαιρούνται και σε υποπρογράμματα. Αλλά δεν δείτε θέμα τεχνικής βοήθειας με εμπειρογνώμονες. Απλά έτσι να δώσουμε ε, κάποια γενική γραμμή και απλά να βοηθήσουμε κράτη να μπουν στον μεταρρυθμιστικό δρόμο. Και διαρωτώ τελικά, ποιο κράτος προαιρετικά θα ζητήσει κάτι τέτοιο και ποια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί, μα ποια κυβέρνηση μπορεί να εμφανιστεί και να πει μόνη της, ξέρετε δεν τα καταφέρνω, παρακαλώ βοηθήστε με Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθήστε με και στείλτε μου ξένους εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, κατά πόσο μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα ερώτηση να την απευθύνουμε και σε κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαδημούλης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρα. Κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Επίτροπε, όπως διαπιστώσατε, υπάρχει και έντονη κριτική στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και πολλά ερωτήματα και μάλιστα από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ομάδων, θα έλεγα από τη μεγάλη πλειοψηφία. Επιτρέψτε μου να επιμείνω, γιατί νομίζω ότι δεν δώσατε επαρκείς απαντήσεις. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές. Πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι επαρκής για να θεραπεύει την αύξηση των ανισοτήτων που έχει προκληθεί και με τη φτώχεια και με την ανεργία και με τις εντυνόμενες κοινωνικές ανισότητες. Επομένως η ανησυχία είναι να μην χαθούν κονδύλια από τις πολιτικές συνοχής με αυτό το νέο εργαλείο που δημιουργείται, αλλά αντίθετα να αυξηθούν τα κονδύλια συνοχής. Ένα πρώτο ερώτημα. Δεσμεύεστε ότι δεν θα χαθούν κονδύλια από τη συνοχή, από τις πολιτικές συνοχής. Δεύτερον, ένα ερώτημα που τέθηκε, άλλες φορές πιο ευθέως, άλλες φορές πιο διπλωματικά, είναι θα πρόκειται για τεχνική βοήθεια ή για πολιτική καθοδήγηση και ε, σε αυτό. Χρειάζεται μια σαφήνεια. Είσαστε οι σοφοί που θεωρείτε το τι είναι το σωστό ή θα βοηθήσετε τις χώρες που χρειάζονται βελτίωση της διοικητικής και της τεχνικής τους ικανότητας για να υλοποιήσουν το σχέδιο που αυτές δημοκρατικά επιλέγουν. Το τρίτο, έχετε υπόψη σας την έκθεση των ελεγκτών για την δουλειά της Tax Force στην Ελλάδα οι ανεξάρτητοι ελεγκτές διεπίστωσαν με μια έκθεση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ελπίζω και εσείς να την έχετε διαβάσει έλλειμμα σχεδιασμού, έλλειμμα λογοδοσίας, έλλειμμα μελέτης επιπτώσεων και μέτρησης των αποτελεσμάτων δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς όπως εσείς σημειώσατε. Για την περίπτωση αυτή. Θα ήθελα να προσθέσω και το τρίτο ερώτημα. Από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά είναι λίγα και που δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια ανάγκη τεχνικής και διοικητικής βοήθειας. Δεν έχει την ίδια ανάγκη η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα με την Γερμανία και την Ολλανδία. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία εσείς θα κάνετε την κατανομή αυτών των κονδυλίων και θα επιλέξετε πού θα δοθεί αυτή η τεχνική βοήθεια έτσι ώστε να πάει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Γιατί πολλές φορές τα κριτήρια που θέτεται με την conditionality ε, την δημοσιονομική οδηγούν ακόμη και τα κονδύλια της συνοχής στις χώρες και τις περιφέρειες που τα έχουν λιγότερο ανάγκη και τα στερούν αυτά τα κονδύλια από χώρες και περιφέρειες και κοινωνικές κατηγορίες που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτά νομίζω ότι υπάρχουν επανειλημμένες εκθέσεις και ψηφίσματα της Επιτροπής Περιφερειών που ασκούν κριτική, που ζητούν αλλαγές. Κλείνω με μια σύντομη αναφορά στη χώρα μου. Η χώρα μου, η Ελλάδα, εφαρμόζει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μεταρρυθμίσεις που αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία. Και αυτό το σημειώνει και το αναγνωρίζει και η Κομισιόν. Στο δε, και αυτό το αναφέρω και σε προηγούμενη συνάδελφο, στο δε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που λύγει η απορροφητικότητα των κονδυλίων στην Ελλάδα και θα ήθελα και τη δική σας επιβεβαίωση Επίτροπη Ταυρόσκης ήταν για την Ελλάδα πρώτη μεταξύ των κρατών μελών, των 28 κρατών μελών. Επομένως, ας μην πυροβολούμε το ασθενοφόρο και ας δούμε πώς θα ενισχύσουμε τις πολιτικές συνοχής εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το τελευταίο ερώτημα. Επίτροπε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Καλώς. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. ως προς ε, τα διάφορα επίπεδα. Το εθνικό με το περιφερειακό. Απαντώ λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και για τις περιφέρειες. Θα πρέπει όμως να υποβληθεί έτοιμα σε εθνικό επίπεδο από το κράτος μέλος. Αν υπάρχει όμως ένα τέτοιο αίτημα, για περιφερειακές μεταρρυθμίσεις, για μεταρρυθμίσεις για ορισμένες πολιτικές που εντάσσονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ε, θα πρέπει το κράτος μέλος να το αιτηθεί. Ε, μας ρωτήσατε για την περίοδο μετά το 2020. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταρτήσει συγκεκριμένες προτάσεις για μετά το 2020. Είναι πρόωρο αυτό το ερώτημα, θεωρώ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποιες πρώτες εμπειρίες και θα μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε πριν καταρτήσουμε πιο συγκεκριμένη πρόταση για το 2020. Στη συνέχεια μου τέθηκε ένα ερώτημα για το πρόγραμμα στήριξης των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και τη τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Το πρόγραμμα αυτό δεν συνεπάγεται αλλαγές στον κανονισμό ΕΣΥΦ και την μακροοικονομική αιρεσιμότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δηλαδή. Δεν ε, θα αλλάξει αυτή η αιρεσιμότητα, οι κανόνες και οι προϋποθέσεις έτσι όπως προβλέπονται στον κανονισμό. Ε, είναι πράγματα που υπάρχουν, έχουν επιβληθεί και ε, ε, τα, συμπεριλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στα εθνικά επιχειρησιακά τους προγράμματα. Τώρα, η σχέση μεταξύ των ειδικών συστάσεων αναχώρα, της τεχνικής βοήθειας και της ευελιξίας. Απαντώ λέγοντας ότι βεβαίως και υπάρχει ευελιξία με την έννοια ότι το κράτος μέλος θα διαλέξει ποιον τομέα χρειάζεται, ε, για ποιον τομέα χρειάζεται τεχνική βοήθεια. δεν είναι ο τομέας προκαθορισμένος από τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Τροποντινά, ε, εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη σε συγκεκριμένη περιφέρεια που ε, συνάδει με τις προτεραιότητες μπορεί το κράτος μέλος να την επιλέξει, να επιλέξει αυτό το τομέα ή αυτό το θέμα και να ζητήσει για αυτό τεχνική βοήθεια και στήριξη. Τώρα, ερωτήσεις που είναι ε, τοποθετήσεις. Έχω ήδη απαντήσει στην προηγούμενο γύρω ερωτήσεων κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έρχεται να ε, υπερκεράσει, λέτε, ή να καπελώσει άλλα προγράμματα. Εγώ θα μιλούσα για συνέργειες. Είναι το θέμα πώς το ερμηνεύει κανείς και ποια αξιολόγηση κάνει. Σίγουρα η πρόταση αυτή είναι ε, εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές. Και προσπαθεί η πρόταση αυτή να ασχοληθεί και να επιλύσει με όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κάθε φορά που χρειάζεται τεχνική βοήθεια προς τα κράτη-μέλη. Και προσπαθεί η πρόταση αυτή ε, να δει πώς διάφορες πολιτικές και διάφοροι τομείς μπορούν να έρθουν και να υποβοηθήσουν. Ως προς τη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα και τις επιδόσεις της Task Force, εγώ ανέφερα αυτό το παράδειγμα και στον προηγούμενο γύρο των ερωτήσεων πράγματι για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων χάρη και με τη στήριξη της Task Force για την Ελλάδα η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ουσιαστικά βελτιώσει την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. και σε άλλους τομείς παρέχεται τεχνική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει το έργο των εμπειρογνωμόνων, των διαφόρων ε, εθνικών εμπειρογνωμόνων από τις διάφορες χώρες. Είτε πρόκειται για την ε, ε, ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, είτε πρόκειται για την ενίσχυση της φόρο πραξιμότητας είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Επομένως η Task Force στην Ελλάδα ασχολείται, η υπηρεσία δηλαδή στήριξης τώρα, ασχολείται με ευρύ πεδίο ε, θεμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014 με 2020. Μας ενδιαφέρει η βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων και η εφαρμογή των ε, προαπαιτούμενων της αιρεσιμότητας εξ άντε εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τέθηκε το ερώτημα ε, του τίτλου 5 η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο τίτλος 5, το πρόγραμμα, ο τομέας 5, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με τη στήριξη στα κράτη-μέλη για τις, για τα, τις διαδροτρωτικές μεταρρυθμίσεις και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί βάσει του τίτλου 5. Ο τίτλος 5 όμως θα χρησιμοποιηθεί για ε, ως κονδύλια για τη διαχείριση του, του προσωπικού. Τώρα, σε σχέση με την ερώτηση για το ποιο κράτος μέλος θα εθελοντικά θα ζητούσε τέτοιου είδους τεχνική βοήθεια. Πρέπει να σας πω ότι ήδη η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιούν εκτεταμένα την τεχνική βοήθεια, αλλά έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο λόγω της ομάδας στήριξης για την Κύπρο και της Task Force για την Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή συζητούμε και με διάφορα άλλα κρατημέλη, τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Συνοψίζω λοιπόν λέγοντας ότι ναι βεβαίως και υπάρχουν κρατημέλη που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και τέθηκε και το αντίθετο ερώτημα. Με βάση ποια κριτήρια θα διαλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις χώρες που θα τύχουν στήριξη. Απαντώ λέγοντας ότι αν η ζήτηση ξεπεράσει την προσφορά, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα κριτήρια, ε, όπως για παράδειγμα το επίγον ε, του προβλήματος αλλά και την ένταση της πρόκλησης, της, ε, την ένταση του προβλήματος στην εκάστοτε χώρα, αναλύοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και τη γενική διοικητική ικανότητα του κράτους μέλους. Βεβαίως θα αξιολογήσουμε και θα βοηθήσουμε πρώτα τα κράτη-μέλη που το χρειάζονται περισσότερο. Τώρα, ως προς το ερώτημα του κατά πόσο οι χώρες θα χάσουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Νομίζω ότι το κατέστησα σαφές στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν αγγίζει τους εθνικούς χρηματοδοτικούς φακέλους των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν χάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα, Εάν πρόκειται για τεχνική βοήθεια ή πολιτική καθοδήγηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τεχνική βοήθεια και ενίοτε μπορεί να φτάσει και σε πολύ ε, βαθύ τεχνικό επίπεδο. Και αυτή την εμπειρία έχουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Τώρα, Μπορεί κανείς, αν αυτό θα στηρίξει τις ε, μεταρρυθμίσεις που ελεύθερα επιλέγουν οι χώρες ε, και ή θα εξαρτάται από τις δημοκρατικές επιλογές και το καθεξής. Η απάντηση είναι ναι, ναι, στο βαθμό που δεν έρχονται οι επιλογές αυτές σε αντίθεση με τις κοινέ προ, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μεγάλη ευελιξία για το ποιες μεταρρυθμίσεις και ποιες, ε, ποιους ε, τομείς ε, πολιτικής μπορούν να διαλέξουν τα κράτη-μέλη για να εντάξουν στο αίτημα τεχνικής τους βοήθειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και Αντιπρόεδρε. Ήταν η πρώτη συνάντησή μας πάνω σε αυτό το θέμα και η πρώτη συζήτηση. Θέλετε να πείτε κάτι. Σε ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων λέει ο κ. και θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Επίτροπο, τον ευχαριστούμε για τις Έχουμε πολύ στριμωγμένο χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε να μεταφραστεί η έκθεσή μας τον Ιούλιο. Δεν αποκλείεται οι εισηγητές βάσει της συζητήσεως να έχουν πιο στοχευμένες ερωτήσεις τις επόμενες ημέρες και θα παρακαλούσα τον κύριο Επίτροπο να είναι διαθέσιμος, να μας βοηθήσει για να πάρουμε τις πληροφορίες. Είσαστε δια... διαθέσιμος. Δεν θέλω να πω ότι είχαμε μια πρώτη συνάντηση και τελείωσε. Πρέπει να μπούμε σε βάθος, όπως είπατε, για την τεχνική βοήθεια. Ίσως πρέπει να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ευχαριστώ. Κυρία Κρέλ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Είναι λοιπόν η πρώτη συνάντηση, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε τις πληροφορίες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Στομπρόσκης, όσον αφορά αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη να παράσχει η αδίποτε συμπληρωματική πληροφορία, ό,τι χρειάζεστε για τις εργασίες σας. Και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία από του θέματος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την τιμότητά σας. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τις εργασίες μας λάβατε τις αποφάσεις των συντονιστών. Αν συμφωνείτε με αυτές, έχουν διανεμηθεί τις θεσινές αποφάσεις. Έχετε κάποια σχόλια? Όχι, εγκρίνονται λοιπόν. Στα διάφορα υπάρχει κάτι? Όχι σήμερα. Σας ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνάντηση Τετάρτη 15 Ιουνίου και 5η 16 Ιουνίου το πρωί και θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και, ε, και εμείς. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.